Καλημέρα συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά λέει ο Πρόεδρος. Ε, ας ξεκινήσουμε παρότι από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά νωρίς ε, για κάποιους συναδέλφους. Λοιπόν, αν δεν έχουμε αντιρρήσει να θεωρήσω ότι έχουμε εγκρίνει το σχέδιο της ημερησίας διατάξεως, στο δεύτερο σημείο, να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της 5ης Φεβρουαρίου, αν δεν έχουμε σχόλια, και εδώ θα θεωρήσω ότι εγκρίναμε Τώρα ανακοινώσεις του Προέδρου, δύο έχω τέτοιες. Καταρχάς, η κυρία Ίσοδος δίπλα στο βήμα θα παραμείνει κλειστή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων για να σεβαστούμε τους ομιλητές. Εάν θέλετε να αποχωρήσετε, να χρησιμοποιήσετε τις πλαϊνές πόρτες, γιατί ενοχλεί η πόρτα αυτή όταν ανοιγοκλίνει διαρκώς. ρακέλα παρακαλώ να αποστείλετε email στους συντονιστές των ομάδων διότι δεν είναι παρόντες όλοι. Θα θυμάστε ότι 21 Ιανουαρίου είχα θέσει το θέμα της εκλογής των ε, των αντιπροέδρων. Είναι 7 ολόκληροι μήνες από τη σύσταση και είμαστε η μόνη επιτροπή στο Κοινοβούλιο που λειτουργεί με έναν μόνο αντιπρόεδρο αυτό υποχρεώνει τον πρόεδρο να έχει υπερβολικά μεγάλη πίεση και φόρτο. Για τους λόγους αυτούς, συμπεριέλαβα στο σχέδιο μερισίες διατάξεως για τις 16 Μαρτίου την εκλογή των υπολοιπωμένων αντιπροέδρων, ώστε επιτέλους, επιτέλους ξαναλέω, να ολοκληρώσουμε. Δεν θα υπάρχει καμία άλλη συζήτηση. Αυτό θα γίνει στις 16 Μαρτίου. Τελεία. Και παύλα. Να ειδοποιήσετε λοιπόν τους συντονιστές και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι αυτή η απόφαση ελήφθη. Πάμε στο σημείο 4. Να καλωσορίσω τον David Beasley, εκτελεστικό διευθυντή του Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφίμων των Ηνωμένων η κυρία Φερέρα είναι εδώ, όχι. Α, είναι, μάλιστα. Ο David Beasley, είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα. Έχουμε μακρόχρονη συνεργασία με το επιστημικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση περιοχών κρίσεων. Η συνεργασία αυτή δεν επιτρέπει μόνο να αυξάνουμε τη δυνατότητά μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε βοήθεια και ενίσχυση, αλλά και σε πολύτιμες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε από την κατάσταση στο πεδίο. Είναι επίκαιρη αυτή η ενημέρωση γιατί θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το πεδίο της συνεργασίας μας. Κύριε Μπίσλε, θέλουμε να μας πείτε πώς αξιολογείται την ανθρωπιστική κατάσταση σε διάφορες δύσκολες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω πρώτα κάποια σχόλια και μετά θα ακούσω τις ερωτήσεις σας για οποιαδήποτε κρίση στον κόσμο. Είμαστε ο μεγαλύτερος οργανισμός ε, τροφίμων στον κόσμο. Το 18, 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν ο προϋπολογισμός όπου μπήκα στο, στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών με μεγάλες αφιβολίες, γιατί είχα, ήμουν καχύποπτος για την μη αποτελεσματικότητα, τώρα είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός του Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφίμων, γιατί είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς οργανισμούς στον πλανήτη Γη, λέει ο ομιλητής. Έχουμε τοποθετήσει κριτήρια αξιολόγησης, ε, ε, έχουμε ποσοτικά κριτήρια για όλα αυτά που κάνουμε, έχουμε στόχους που τους καλύπτουμε, αλλά δυστυχώς οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται ταχαίως στον κόσμο. Το 19 ήταν πολύ πολύ κακή χρονιά και για να είμαι ειλικρινής το 20 φέτος θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Αν δείτε τις διάφορες κρίσεις, ο προϋπολογισμός σε λίγα χρόνια από 4,5 δις πήγε σε περί τα 8,5 σχεδόν. Και καθότι διάφοροι άλλοι προϋπολογισμοί περικόπτονται, ο δικός μας αυξάνεται, διότι βρισκόμαστε στην πιο στρατηγική θέση ώστε να μοχλεύσουμε τη συνεισφορά των φορολογουμένων σε οποιαδήποτε χώρα, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, παντού στον κόσμο, γιατί όλοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν καλύτερα την απτή και συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των τροφίμων και της επιστηστικής ασφάλειας. Εξού και πέρυσι είχε ψήφισμα ο ΙΕ, όπου εξηγούσε ότι χωρίς επιστηστική ασφάλεια δεν υπάρχει καμία άλλη ασφάλεια. Και παρότι ο πληθυσμός της γης έφτασε από το 1 και κάτι στα 7,2 δις, η ένδια και η ασυτεία μειώθηκε δραστικά. 95% ήταν πριν από κάποια χρόνια η απόλυτη ένδυα στον κόσμο, οικοδομήσαμε συστήματα, την πήγαμε στο 85, έχουμε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, αλλά Παρότι λοιπόν κάτω του 10% είναι η απόλυτη φτώχεια στον κόσμο, αυτό πριν από κάποια χρονιά ήταν 770 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Σήμερα είναι 820 εκατομμύρια αυτοί που πεινούν. Και επομένω, ο δείκτης της πείνας, αν θέλετε, αυξάνεται. Και μάλιστα της απόλυτης ασυτείας. Από 80 εκατομμύρια πήγε στα 115 εκατομμύρια. Άνθρωποι δηλαδή που θα κάνουν ό,τι μπορούν για να επιβιώσουν. Και αυτό μπορώ να σας πω από το πρόγραμμα τροφίμων, όταν χρειάζεται να θρέψει κανείς 85-90 εκατομμύρια οποιοδήποτε χρονική στιγμή του έτους, αν το σκεφτείτε αυτό για μια περίοδο 2-3 ετών συνεχομένη, τότε αντιλαμβάνεστε ότι γνωρίζετε τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή. Και ξέρουμε για την Μπόκο Χαράμ, για την Αλκάιντα, για την ISIS. Βλέπουμε τους πρόσφυγες, τις μετακινήσεις πληθυσμών, όλα αυτά. Βλέπουμε όλους αυτούς που είναι ευάλωτους, ακάλυπτους, σε κρίση, σε εμπόλεμες ζώνες, σε συγκρούσεις, σε οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση. Τώρα, αυτό που προκαλεί την αύξηση της αστείας και της πείνας είναι οι κρίσεις, οι ε, εμπόλεμες κρίσεις, Συρία, Σουδάν, Νιγηρία, όπου θέλετε. Αλλά βέβαια και οι ακρότητες ε, του κλίματος. Με κυκλώνες, τυφώνες, η αποσταθεροποίηση που έχει συμβεί λόγω ξηρασίας ή λόγω πλημμυρών. Και όταν μιλάω με τους ε, συντηρητικούς φίλους μου στο, στις Ηνωμένε Πολιτείε, αν δείτε το ποστό βροχόπτωσης σε κάποια χώρα που δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, και το συγκρίνετε με, την, με το δυναμικό κάθε εποχής πόσες πλημμύρες έχουμε π.χ. αντιλαμβάνεται κανείς πόσα εκατομμύρια στον κόσμο και ιδιαίτερα στο Σαχέλ έχουν αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Οπότε μαζί με τις συγκρούσεις, το κλίμα και αν το συνδυάσετε αυτά με τις εξτρεμιστικές ομάδες, την ISIS που συνεργάζεται με την Boko Haram στο Σαχέλ, για παράδειγμα, αντιλαμβανάστε γιατί έχουν αποσταθεροποιηθεί τα πράγματα. Τώρα, αν με ρωτούσε κάποιο πριν από δύο χρόνια ποια είναι τα καλά νέα, θα του έλεγα ότι αποκλείεται το Σουδάν να είναι το καλό μα παράδειγμα στην Αφρική. Αλλά με όλε τι προσπάθειε που έχουμε κάνει στου τελευταίου έξι μήνε, το Σουδάν βρίσκεται σε μια μαγική καμπή της ιστορίας του. Είμαι αισιόδοξο, αλλά και ανησυχώ αισιοδοξώ διότι πιστεύω ότι η ηγεσία έχει μια κατεύθυνση, θέλει να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε συζητήσει με την ηγεσία του Σουδάν, με τους αντάρτες στο Νότιο Σουδάν και είναι απίστευτη η συνεργασία που έχει λάβει η χώρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού των ενόπλων ανταρτών. Αλλά ανησυχώ επίσης γιατί δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η διεθνή κοινότητα κινείται αρκετά γρήγορα ώστε να σταθεροποιήσει αυτήν την πολύ εύθραυστη ισορροπία. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, γρήγορα, τότε μπορεί να επανέλθει η κατάσταση σε ακόμα χειρότερο σημείο από αυτό που ήταν πριν. Και τότε θα έχουμε χρησιμοποιήσει για όλη τη Σομαλία, την Αιθιοπία, όλη την περιοχή ένα στο σημείο. Η Σομαλία προσπαθεί. Η Μπουρκίνα Φάσο έχει αποσταθεροποιηθεί επίσης. Το Μαλί, ο Νίγηρας. Και καθότι προσθέτουμε, καθώς προσθέτουμε κομμάτια στο πάζελ αυτό, στο Σαχέλ, μόνο στους τελευταίους μήνες χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Η μισή από αυτούς άμαχοι Χιλιάδες σχολεία κλείνουν, νοσοκομεία, κλινικές, λόγω των ενόπλων ομάδων αυτών. Διάβαζα τη, τις άλλη, κάποια προηγούμενη μέρα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, αποσύρονται από το Σαχέλ. Σήκουσα το τηλέφωνο αμέσω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή ε, Προπολογισμού και του είπα αμυντικών θεμάτων, του είπα αν τα κάνετε αυτά θα είναι καταστροφικά. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο για την ασφάλεια την στρατιωτική δηλαδή, αλλά αν δεν έχουμε τέτοια συνεργασία, το Σαχέλ θα αποσταθεροποιηθεί πλήρως. Τώρα ακούμε πολλή προπαγάνδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χρηματοδότηση, την πολυμέρεια κτλ. Και αυτό το λέω και από τις δύο μεριές της λεωφόρου Πενσιλβένια. Όταν έφτασα εγώ, είχαμε όπως σας έλεγα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό. Σήμερα ο προπολογισμό από τις ΗΠΑ είναι 3,4 δισεκατομμύρια. Το λέω διότι το μήνυμα που μου στέλνει και ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι του Κοινοβουλίου και στις δύο αίθουσες είναι ότι καταλαβαίνουμε τη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνουμε την κατάσταση στο Σαχέλ, στη Βόρεια Αφρική, παντού ε, και εγώ του έχω πει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλες ευρωπαϊκέ χώρες και αυτοί εντείνουν τι προσπάθειές τους. Επομένως σας ευχαριστώ. Πέρυσι ήσασταν στα περίπου 600 εκατομμύρια και προβλέπεστε για το 19 στα 2,5 δις. Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι η διεθνή κοινότητα εντείνει τις προσπάθειές της. Τα κακά νέα, και δεν μου αρέσει που το λέω, είναι ότι αυτά δεν φτάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες στον κόσμο θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες, ακόμα περισσότερες από όλη την προσπάθεια που έχει γίνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί προκειμένου να σταθεροποιηθούν αυτές οι αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσεις που ποτέ δεν είχαμε δει στο παρελθόν, εάν δεν εντείνουμε τις προσπάθειές μας θα υπάρξει καταστροφή και για να αναφερθώ και στις, ε, στα αίτια του προβλήματος στη Συρία. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τη Συρία θα χρειαζόμαστε 50 σεν την ημέρα. Και αυτό είναι διπλό κόστος από το κανονικό διότι έχουμε πόλεμη ζώνη, έχουμε πόλεμο. Ας πάρουμε ένα Σύριο που ε, ζούσε στη Δαμασκό, αν ήταν στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο, τότε θα ήταν 50 με 100 ευρώ την ημέρα το κόστος, η πρόβλεψη. Δεν θέλουν να φύγουν. Όταν κανείς ρωτάει πρόσφυγες, ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, θα μετακινηθούν τρεις και τέσσερις φορές μέσα στη χώρα προτού εγκαταλείψουν τη χώρα. Είτε μιλάμε για Τσάντ, είτε για τον Νίγερα, είτε για την Πορκίνα Φάσο, οπουδήποτε. Δεν επιθυμούν να φύγουν. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης, του προσφυγικού, αν δούμε τα η Ιδάλλως οι συνέπειες θα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρές. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κρίση με τις ακρίδες, τον κορονοϊό ή την Ιντλίμ, στη Συρία. Ε, πολλά προβλήματα. Εμείς, όπως λέω συχνά, χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα ως όπλο υπέρ της ειρήνης για να ειρηνοποιήσουμε περιοχές, να αντιμετωπίσουμε εξτρεμιστικές ομάδες και γι' αυτό η υποστήριξή σας είναι κρίσιμη. Μπορώ να συνεχίσω όση, όση ώρα θέλετε και μπορώ να πάω σε λεπτομέρειες για όλες αυτές τις κρίσεις. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ερωτήσει για την Ιεμένη, για τη Συρία, τη Βενεζουέλα, τη Βόρειο Κορέα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα το πρωί, αλλά πρόεδρε, δεν ξέρω, President Chairman τι πρέπει να λέω κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να επισκεφθείτε και την έδρα μας στη Ρώμη για να δείτε τις χαρτογραφίσεις που έχουμε, τις απεικονίσεις για τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα λαθρεμπόριο δηλαδή, τις τρομοκρατικές ομάδες, τις ένοπλες ομάδες, τι αντιμετωπίζει δηλαδή ο κόσμος στις χώρες του. Και να σας πω και μια μικρή ιστορία. Εμείς παραδοσιακά χειριζόμασταν μόνο αγαθά. Τώρα είναι διαφορετική η κατάσταση. Διαφορετικό το παιχνίδι. Στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80 είχαμε ανθρωπιστικά παιδεία και ε, αναπτυξιακά παιδεία. Τώρα πρέπει, πρέπει να συνδυάζονται όλα αυτά και να δίνουμε στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία. Γιατί δεν είναι αρκεί μια απλή προσέγγιση όπως ήταν πριν από 30 χρόνια ή 40. Χρειάζεται ευελιξία με την ανθρωπιστική βοήθεια για να επιτύχουμε στόχους. Π.χ. στο Σαχέλ πήραμε ανθρωπιστικά κονδύλια, δουλέψαμε με δικαιούχου ούτε έναν δεν βρήκα που να μην ήθελε να επιβιώσει. Παρότι μπορεί να μην ήθελε βοήθεια. Δηλαδή, να σας δώσουμε τρόφιμα, αλλά να δούμε πώς είναι υγιές. Πώς έχει η κατάσταση στην καλλιέργεια έχουμε περί τη μισή επιφάνεια της χώρας του Βελγίου έχουμε αναδιαρθρώσει με υδροδοτικά έργα, με άλλα έργα για τις καλλιέργειες. Εγώ μιλούσα με μια γυναίκα, μιλούμε για περιοχές τώρα όπου οι γυναίκες είναι καταπιασμένες. Εμείς δουλεύουμε και με τις γυναίκες και με τους άνδρες και είναι απίστευτο όταν βλέπει κανείς τις γυναίκες που αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, δουλεύουν, συνεργάζονται με το δικό μας πρόγραμμα και μας λένε πλέον δεν μπορώ απλώς να θρέψω την οικογένειά μου αλλά πουλάω και στην αγορά, την τοπική. Δηλαδή με αυτή την αναδιάρθρωση των γεών μετά πάμε σε άλλα σχολικά ε, προγράμματα για τα παιδιά και τότε αυτή η ακραία ανάγκη κατέρχεται εντυπωσιακά. Κατέρχεται εντυπωσιακά επίσης ο προσελητισμός από τις τρομοκρατικές ομάδες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών κατέρχονται εντυπωσιακά. Δηλαδή μπορεί να τα δει κανείς όλα αυτά. Είναι πολύ φθηνότερο να αντιμετωπίσουμε τα βασικά αιτία παρά τα συμπτώματα. Και κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να ανησυχεί για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να σας δώσω μια έτσι εικόνα, σύνοψη. Παρακαλώ Πρόεδρε, όποια ερώτηση έχετε στη διάθεσή σας. Thank you. Ευχαριστούμε David Beasley για τις εισηγητικές αυτές παρατηρήσεις. Συνάδελφοι, έχουμε περίπου μισή ώρα για ανταλλαγή απόψεων με τον προσκεκλημένο μας, τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Πιστιστικού Προγράμματος. Μια παρατήρηση να κάνω. Μιλήσατε για το Σουδάν και ήταν ενδιαφέρον αυτό, διότι θα κάνουμε μια επίσκεψη στις αρχές Απριλίου στο Σουδάν και στην ε, Αιθιοπία ως Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα χώρα αυτή και ήταν εξαιρετικά αισιόδοξα τα όσα μας είπατε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, σε σύγκριση με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τουλάχιστον πολλές φορές. Να σας δώσω το λόγο, παρακαλώ έως τρία λεπτά ο καθένας, πρώτος ομιλητή εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριο Κουμπίλιου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εντυπωσιακά τα όσα κάνατε. Έχω κάποιες απλές ερωτήσεις. Είπατε ότι ο προπολογισμό σας αυξήθηκε από 4,5 σε 8,5 δις. Τι προπολογισμό όμως θα θέλατε να έχετε. Δεύτερη ερώτηση για την κλιματική αλλαγή. Ποιε είναι οι προβλέψεις σας. Θέλω να πω, αν συμφωνήσουμε ότι οι θερμοκρασίε αυξάνονται και ότι η κλιματική αλλαγή προχωράει, αυτό θα σημαίνει ότι θα ενισχυθούν και τα προβλήματα στην Αφρική. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε 10 χρόνια. Έχετε προβλέψεις, εκτιμήσει, τι προπολογισμό θα χρειαστείτε για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Go one on one? Okay, fine. Απαντήστε παρακαλώ κύριε Μπίσλη. Κύριε Πρωθυπουργέ, 12 εκατομμύρια θα έλεγα. Με, δις, δις, συγγνώμη. Δις εκατομμύρια. Αλλά πρόκειται για έκτακτη βοήθεια. Για να υπάρχει πραγματική επιστηστική ασφάλεια, για να είναι βιώσιμη, χρειαζόμαστε υψηλότερο προϋπολογισμό και βραχυπρόθεσμα. Γιατί όσον αφορά τα στρατηγικά προγράμματα, εγώ ε, θέλω να υπάρχει μια ε, μακροχρόνια στρατηγική και να μην υπάρχουν συγκεκριμένες διακυμάνσεις του προϋπολογισμού ευξήσεις, εκτός αν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη, κρίση, όπως ε, ένας τυφώνας για παράδειγμα ή κάτι τέτοια. 12 δις θα θέλαμε. Κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορεί κανείς να συζητά ε, επί μακρόν τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή δεν είναι δική μου υπόθεση να δώσω την οριστική απάντηση. Εγώ μπορώ να σας πω τι γίνεται επί τόπου. Εμείς περιμένουμε τα επόμενα 20 με 30 χρόνια να υπάρξουν 200 εκατομμύρια εκτοπισθέντες, εσωτερικά εκτοπισθέντες ή γενικά εκτοπισθέντες, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 95 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ε, πληγεί δραματικά από την ε, κλιματική αλλαγή. 29 εκατομμύρια άνθρωποι ήδη αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας λόγω της ε, κλιματικής αλλαγής. Αυτό που εμείς θα θέλαμε να κάνουμε είναι να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Αφγανιστάν. Παραδοσιακά ε, πηγαίναμε τρόφιμα και τα παραδίδαμε στους ανθρώπους εκεί. Στην Μάζορα Αλσίφ, για παράδειγμα, γιατί γίνονταν πλημμύρε, για παράδειγμα, και κατέστρεφαν τι καλλιέργειε. Τι κάναμε εμεί λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει. Με τη ΣΥΠΑ που ήταν ο δωρητή. Είπαμε, αντί να φέρουμε τρόφιμα απ' έξω, δώστε μα χρήματα να συναντηθούμε με του γεωργού, με του αγρότε εκεί, στι πιο έφορε πεδιάδε του Αφγανιστάν και θα θα κάνουμε τα εξή. Θα του κάνουμε μια συμφωνία ότι θα αγοράσουμε αυτέ τι ποσότητε σε αυτή την τιμή για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να προσλάβουν κόσμο, να αγοράσουν εξοπλισμό και αυτό. Πήραμε δηλαδή τα ίδια χρήματα, αντί να του δώσουμε τρόφιμα, τα μετατρέψαμε σε οικονομική βοήθεια για του ανθρώπου στους Αφγανιστάν. Από εκεί και πέρα πήραμε τα τρόφιμα στη Μάζιρ Σαρίφ και του είπαμε θα σας δώσουμε αυτά τα τρόφιμα, αλλά γιατί, για να αποκαταστήσουμε το τοπίο, ώστε όταν υπάρχουν πλημμύρες από τις βροχοπτώσεις θα υπάρχουν συστήματα ε, διαχείρισης των υδάτων για να μην καταστρέφονται οι καλλιέργειές σας. Και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ρώτησα πρόσφατα έναν γεωργό τέτοιο που είχαμε συνεργαστεί και του είπα πώς άλλαξε η ζωή σου. Και ήταν τόσο περήφανος και μου είπε ότι τα παιδιά μας σταμάτησαν να φεύγουν από τα σπίτια, από τις, από, από τις πόλεις μας. Δεν πηγαίνουν στους Ταλιμπάν ή στις ε, αντικυβερνητικές ε, αντάρτικες ομάδες. Γιατί τώρα πια το νερό ε, εκτρέπεται αλλού και δεν καταστρέφει τις καλλιέργειες μας και τώρα πια μπορούμε να μείνουμε εδώ. Αυτή είναι η διαφορά. Πηγαίνουμε σε περιοχές, αποκαθιστούμε τις ε, καλλιεργούμενες εκτάσεις και φέτος μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες ε, φυτέψαμε 5 έως 6 δισεκατομμύρια δέντρα, μόνο πέρσι εκατοντάδες εκατομμύρια, αποκαταστήσαμε καλλιεργήσιμες εκτόσεις, χτίσαμε 15.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου που βοηθά την μεταφορά τροφίμων, τις εμπορικές διαδρομές, διάβλους, κανάλια, ε, παιδιάδες αποστράγγισης και έτσι αποκαθιστούμε και αντιμετωπίζουμε τους λόγους που ανεξάρτητα μάλλον από τους ποιοι είναι οι λόγοι που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, εμείς βοηθούμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα για να μπορούν να επιβιώσουν και είναι πραγματικά μια τεράστια διαφορά που έχουμε επιτύχει επιτόπου. Με, σε σύγκριση με μόλις πριν από λίγα χρόνια, την κατάσταση που επικρατούσε πριν από λίγα χρόνια. Και δεν μιλώ καν για Αφρική, για άλλε περιοχέ. Σα μιλώ μόνο για αυτό το παράδειγμα. Υπάρχει ένα σχεδιασμό τεράστιο, οργιώδη για το τι κάνουμε και ζητούμε από, τα, από το Υπουργείο να μα δώσουν περισσότερα κονδύλια για να μπορούμε να ε, τροποποιούμε και τι διάφορε παρεμβάσει μα. Πάντως είναι πολύ πιο πολυσχηδή η παρέμβασή μα σε σχέση με το τι κάναμε πριν από μερικά χρόνια. Ο κύριο Σιμοσέβιτ από του σοσιαλιστέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το κοινοβούλιο αυτό ε, σας επισκέφτηκε στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο. Και πρέπει να πω ότι οι πληροφορίε που μα έδωσε ο αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για το ίδιο θέμα ήταν από τι πιο εντυπωσιακέ που ακούσαμε στην επίσκεψή μας στον ΟΗΕ. Και θέλω να σας πω ότι και αυτά που μας παρουσιάσατε και εσείς σήμερα είναι και ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά και νομίζω ότι η δραστηριότητα του ΟΗΕ σε αυτόν τον, σε αυτόν τον τομέα πραγματικά ε, ε, χαίρει της εκτίμησής μας. Είπατε ότι σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις αντί για την παραδοσιακή βοήθεια και αρρωγή μέσω της παροχής τροφίμων αποφασίζεται να υποστηρίζεται λύσεις ε, για την αντιμετώπιση της πείνας με χρήματα. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγετε το ένα ή το άλλο πρόγραμμα. Επίσης, αναφερθήκατε στη Βόρεια Κορέα ως χώρα που βοηθάτε. με. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βόρεια Κορέα και τη βοήθεια που παρέχετε στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Μπίζλι, ναι. Όταν ε, ανέλαβα τα καθήκοντά μου πριν από τρία χρόνια, είχα πολλέ επιφυλάξει σχετικά με τα μετρητά χρήματα, γιατί μπορεί να καταλήξουν στου λάθο ανθρώπου και δεν το θέλει αυτό. Ταυτόχρονα όμως ε, ε, εξηγούμε με τι ομάδε μα ποιες, πότε χρησιμοποιούμε πότε, και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα χρήματα στους δωρητές μας. Ε, εγώ όταν έφτασα είχαμε 250 εκατομμύρια ε, δολάρια. Σήμερα οι σχετικές δαπάνες μας σε μετρητά ήταν 2,1 δις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ιεμένη, όπου οι Χούτι ε, εκτρέπουν την, την παροχή τροφίμων, στρεβλώνουν με διάφορους τρόπους την αγορά τροφίμων για να ανεβαίνουν οι τιμές, όπως γίνεται και στην στην Συρία. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά όταν πηγαίνουμε σε συγκεκριμένε περιοχέ και δεν χρησιμοποιούμε εμπορεύματα, αλλά χρησιμοποιούμε μετρητά και έχουμε βιομετρικά δεδομένα ώστε να εξασφαλίζουμε ότι ο κάθε δικαιούχο είναι ο πραγματικό δικαιούχο, αυτό που παίρνει τα χρήματα είναι αυτό που τα δικαιούται. Με αυτόν τον τρόπο, εμεί βοηθούμε 2,8 εκατομμύρια από, ε, ιεμένους από τους, ε, από τους 30. Σημαίνει ότι αν πάμε με πρόγραμμα μετρητών χρημάτων θα δοθούν κίνητρα στην οικονομία με, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές των τροφίμων συνολικά. Γι' αυτό και εμείς καλούμε κυβερνήσεις και η ΙΠΑ συνήθως παραδοσιακά δίνανε μόνο τρόφιμα, μόνο εμπορεύματα δίνανε μέχρι από πέντε χρόνια. Από 3,5 δις που δίνουν ε, πλέον οι ΙΠΑ, το 50-60% είναι μετρητά χρήματα. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Να μας δίνετε χρήματα ώστε να μπορούμε να τα ανακατευθύνουμε εμείς εκεί που πρέπει. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία με αυτή την Ζητάμε από τις κυβερνήσεις να μας δίνουν χρήματα. Γιατί όταν υπάρχει έλλειψη υποστήριξης προφανώς θα πάρεις ό,τι, ό,τι σου δώσουν. Όμως με τα χρήματα μπορούμε και να αγοράζουμε τροφήματα. Γιατί σε κάποιες περιοχές όπως στη Συρία ή αλλού δεν υπάρχει αγορά. Δεν μπορεί κανείς να βρει τρόφιμα στην αγορά. Οπότε εκεί ναι πρέπει να πας τρόφιμα, να μεταφέρεις τρόφιμα. Αλλά αν υπάρχει αγορά η οποία είναι σχετικά σταθερή και μπορείς να χρησιμοποιήσεις βιομετρικά δεδομένα ώστε να αποφεύγεις απάτες κτλ, τότε ναι μπορούμε να δίνουμε και μετρητά χρήματα. Βιομετρικά δεδομένα και ψηφιοποίηση από τότε που, τα έχουμε φτάσει, από τότε που έφτασα εγώ έχουμε αρχίσει μια διαδικασία ψηφιοποίησης και πλέον έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει 50 εκατομμύρια δικαιούχους τα βιομετρικά του δεδομένα και αυτό μας δίνει μεγάλη ευελιξία στις δράσεις μας. Και χρησιμοποιούμε βεβαίω και εμπορεύματα, τρίβματα, ε, βιομετρικά δεδομένα μάλλον, και για, και για τα χρήματα και για τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα όταν δίνουμε. Αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικά εύρωστα τα συστήματά μας όταν έχουμε βιομετρικά δεδομένα μαζί με την ψηφιοποίηση και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν παραμέτρους που χρησιμοποιούμε σε όλα, σε σε όλα τα κράτη. Υπάρχει μια ολόκληρη διάρθρωση βεβαίω, αλλά είναι μια συζήτηση που γίνεται σε πολλέ χώρε. Στο Λίβανο, για παράδειγμα. Αν πάμε τρόφιμα στο Λίβανο, ε, και ξέρετε ότι εμείς ε, ε, σητίζουμε ένα εκατομμύριο ανθρώπους στο Λίβανο. Αν σηκωθούμε και φύγουμε, τότε οι επιπτώσεις οι οικονομικές θα είναι καταστροφικές. Όμως έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα μεταφοράς χρημάτων. Αν πάμε εκεί εμπορεύματα, τότε προφανώς θα καταστρέψουμε την αγορά, γιατί θα καταρρεύσουν οι τιμές. Έχουμε λοιπόν οικονομολόγους, οι οποίοι παίρνουν υπόψη τους γεωργικά δεδομένα και άλλα δεδομένα, για να δούμε ποια είναι η πλέον στρατηγική επένδυση και μετά το συζητούμε αυτό με τον δωρητή που θέλει να χρηματοδοτήσει ό,τι του προτείνουμε εμεί, εν πάση το συζητάμε. Στο Λίβανο, για παράδειγμα, έχουμε προσδιορίσει πάνω από 500 μικρά καταστήματα. Και ένας Σύριος πρόσφυγας, για παράδειγμα, μπορεί να πάει με μια ε, μικρή καρτούλα, σαν πιστοτική, για παράδειγμα, που μπορεί να περιλαμβάνει και τα βιομετρικά του δεδομένα και μπορεί να αγοράσει συγκεκριμένα ε, προϊόντα από αυτό το κατάστημα. Έτσι όμως σταθεροποιείται και η οικονομία του Λιβάνου και ταυτόχρονα δίνουμε και μια μεγαλύτερη πολυμορφία, ελευθερία στον πρόσφυγα για να μπορεί να έχει μια όσο το δυνατόν πιο κανονική και ομαλή ζωή. Και θα μπορούσα να σας δώσω και άλλα παράδειγμα, αλλά έτσι ενδεικτικά. Α, Βόρεια Κορέα, ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Για τη Βόρεια Κορέα να σας πω τα εξής. Είχαμε διαπραγματευτεί με την Βόρεια Κορέα και με κάποιους μεγάλους δωρητές. Πλέον παρέχουμε βοήθεια σε 500.000 έως 1 εκατομμύριο ανθρώπους στη Βόρεια Κορέα. Κάναμε και μια τελευταία αξιολόγηση το καλοκαίρι το φθινόπωρο. Η Βόρεια Κορέα ανησυχεί πάρα πολύ για την κατάσταση που επικρατεί. Βρισκόμαστε σε επαφές μαζί τους. Ε, με ουδετερότητα και ανεξαρτησία γιατί οι δωρητές είχαν μεγάλη ανησυχία ότι οι προοριζόμενοι δικαιούχοι ε, θα λάμβαναν ε, τρόφιμα αντί για να μην καταλήξουν τα χρήματα που δίνουν στο στρατό της Βόρειας Κορέας Κάναμε λοιπόν πολύ λεπτομερείς ε, διαπραγματεύσεις. Σχεδόν είχαμε φτάσει στη σύναψη και τελικά ήρθε η Κίνα και έδωσε εκατο... εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ε, ε, τόνους εμπορεύματα, τρόφιμα και φυσικά ο ρόλος μας εκεί σταμάτησε κατευθείαν. Ο ρόλος μας είναι ο εξή. Φυσικά η κατάσταση χάρη στην βοήθεια της ε, Κίνας βελτιώθηκε. Δεν ξέρουμε όμως πού ακριβώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση για το πού βρισκόμαστε. Φυσικά και ο κορονοϊός έχει διαταράξει τις ομαλές ροές εμπορευμάτων και υπηρεσιών βεβαίω σε ολόκληρη την, την ευρύτερη περιοχή. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση αξιολόγησης για το πού βρισκόμαστε. η Νότια Κορέα έχει ε, δώσει επίσης ε, μεγάλη βοήθεια. 50.000 τόνους τρόφιμα θέλει να δώσει η Νότια Κορέα στη Βόρεια Κορέα. Τα αρνείται βεβαίως η ε, Βόρεια Κορέα. Υπάρχουν και άλλες χωρές, η Ρωσία, η Ελβετία έχουν δώσει εκατομμύρια, τα έχουν θέσει στη διάθεσή μας αν θέλετε. Ε, αυτή είναι η κατάσταση μετά την ε, τελευταία παρέμβαση των ε, Κινέζων που παρέσχουν αυτή την βοήθεια στην Βόρεια Κορέα. Ευχαριστώ. Δεν έχω έτοιμα από την ομάδα Ρινιού. Περνάω όμω στου πράσινου ο κύριος Λάγκενσίγκερ. Κυρία Λάγκενσίγκερ. Ευχαριστώ. Στα γερμανικά θα μιλήσω, οπότε σα παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ θέλω να σταθώ στη Συρία. Ο πόλεμος στη Συρία είναι ένας πόλεμος ε, διαντιπροσώπων. Δεν είναι εμφύλιος πόλεμος. Είναι ένας ε, πόλεμος ο οποίος έχει προκαλέσει 900.000 πρόσφυγες σε μεγάλο βαθμό παιδιά. Εσείς περιγράψατε το idlib. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διερμηνία. Ah, there's no trans... Oh, okay. I didn't know. <laughs> I restart. Να ξαναξεκινήσω. Test, test, 2, 3. Herzlichen Dank. Could the English interpreter say something? No. Okay. No. No. Good. Sorry. Ωραία, υπήρξε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο, αλλά νομίζουμε ότι λύθηκε. Now it's working. Now it's fine. For everyone? Okay. Ich beginne dann noch einmal. Ωραία, ξαναξεκινάω. Ο πόλεμος ε, της Συρίας, όπως έλεγα, είναι πόλεμος διαντιπροσώπων. αντιπροσώπων. Δεν είναι εμφύλιος πόλεμος. Μιλάμε για 900.000 πρόσφυγες, 60% είναι παιδιά και έφηβοι που δεν εμφανίζονται πουθενά, ούτε στατιστικές. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι στην, στο Ιγκλίπ, που είναι μια ζώνη αποκλιμάκωσης, το να φύγει κανείς από εκεί είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορεί κανείς να κάνει στον πλανήτη Γη. Εσείς ως ε, μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές ε, βοήθειας, ε, οργανώσεις βοήθειας. Είπατε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωπο στηρίζεται και επισητίζεται και από την χώρα αυτή καταφθάνουν βεβαίως και εκατομμύρια πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες και αλλού. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι η Τουρκία παρά τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, έχει αρχίσει να ε, κατασκευάζει εστίες επισυριακού εδάφους και μάλιστα και με την ανοχή της γερμανικής κυβέρνησης. Είναι πραγματικά κατά τη γνώμη σας η μόνη ρεαλιστική λύση για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Ποιε είναι συγκεκριμένα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε επί τόπου. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα διατυπώνεται το αίτημα δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων. Είναι εφικτό να δημιουργηθούν τέτοιοι διάδρομοι ανθρωπιστικής βοήθειας και ποιες παράμετροι θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. Με απότερο σκοπό βεβαίως τον τερματισμό της πολεμικής ε, σύγκρουσης. Ο, η, ε, ε, είπατε εκπρόσωπες για την εξωτερική πολιτική ε, <clears throat> έχει ε, περιγράψει τις κόκκινες ε, γραμμές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει βοήθεια για την οικοδόμηση αυτών των οικειών επισυριακού εδάφους. Ποια είναι η δική σας άποψη από οργανωτικής άποψης, από άποψη επιμελητίας, τι χρειάζεστε. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε δύο ομιλητές και μετά θα δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Μπίσλι για να ε, ολοκληρώσει. Ο κύριος, η κυρία Φωτίγκα. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντή που έχετε μοιραστεί τις απόψεις σας μαζί μας που ήρθατε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρακαλώ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες σας σε όλους τους συνεργάτες σας. Μας εντυπωσιάζει πραγματικά ε, αυτό που πετυχαίνετε στο πιστιστικό πρόγραμμα. Επειδή, επειδή ξέρουμε και το ιστορικό και προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν, πιστεύω ότι οι τρέχουσες δραστηριότητες είναι πραγματικά εντυπωσιακέ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε προηγούμενη ερώτηση που έχει τεθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους παίκτες που εμπλέκονται στη Συρία σήμερα. Πώς βλέπετε τη δυνατότητα σήμερα να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά σε κρίσεις όπως αυτές που διαφαίνονται στο Ιντλίπ, όπου χρειάζεται να παρασχεθούν πολλαπλά αγαθά και όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και θέρμανση και ανταπόκριση σε ανθρωπιστική κρίση. Ε, υπάρχει υποσυτισμός ε, που αναπτύσσεται ε, εκεί, καθώς και η ανάπτυξη επιδημιών. Από την άλλη πλευρά στην Αφρική έχουμε μια μεγάλη εμπλοκή της Κίνας Πώς βλέπετε εσείς τις δικές σας δραστηριότητες σε σχέση με αυτές τις κρίσεις και σε, ειδικά σε περίπτωση ε, διάδοσης επιδημιών στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επίσης. Πώς αντιμετωπίζετε, έχετε ειδικά προγράμματα για να αντιμετωπίσετε, για παράδειγμα, παιδιά που πάσχουν από σοβαρές περιπτώσεις υποσυτισμού ε, εκτός από τα μικρής κλίμακας προγράμματα στο Ανατολικό Κονγκό, ε, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να υπάρχουν, γιατί προποθέτει διαφορετικού τύπου σύντησης και όχι απλά παροχή τροφής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τελευταίος ο μιλητής Chris Peters. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς τον Διευθυντή για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί τώρα και θα επιτελέσει και στο μέλλον. Μια επίκαιρη ερώτηση. Αντιληφθήκα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη Σομαλία, Αιθιοπία και Έννοια με την, ε, το πρόβλημα με τις ακρίβες. 15 εκατομμύρια κρίδες ε, προς ε, ε, επιτίθενται στην περιοχή κάθε μέρα. Και το πρόβλημα είναι, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε, είναι μέρος της των θεμάτων της κλιματικής αλλαγής. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιου είδους μαζικές καταστροφές γιατί καταλαβαίνω ότι πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τροφή. Σας ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν. Ε, τελικός γύρος και θα κλείσουμε στις 10 παρα 5. Συρία πρώτα. Η Συρία αυτή τη στιγμή ε, εκεί ξεδιπλώνεται το θέμα. Στην Συρία ε, στηρίζουμε 4,5 εκατομμύρια. Το 2017-2018, λόγω των δραστηριοτήτων μας, ε, είδαμε τις τιμές των εμπορμάτων να μειώνονται ε, σε ένα έθνος 22 εκατομμύριων. Αλλά λόγω της σύγκρουσης και της επιδείνωσης της κατάστασης, οι τιμές των αγαθών αυξάνονται και για την υπόλοιπη χώρα που δημιουργεί προβλήματα εκεί. Η πρόσβασή μας ε, στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά, ανεξαρτήτως της πολιτικής, όμως στο Ιντλίπ υπάρχει κρίση και ε, αλλάζουν τα πράγματα με την ώρα, όχι με την μέρα οι επιχειρήσεις αλλάζουν την κατάσταση με την ώρα. Βλέπετε το χάρτη αυτό. Είναι ένας χάρτης της Συρίας και της Τουρκίας. Ε, με πορτοκαλί βλέπετε τις περιοχές υπό τον έλεγχο της Ιρακής κυβέρνησης. Μετά έχουμε την, ε, τις, περιοχές που ελέγχονται από την Τουρκία και από τους Αντάρτες και έχουμε τις μεθοριακέ γραμμές. Εκεί ε, πρέπει εμείς να περάσουμε με τις παροχές τροφίμων, θα πρέπει να περάσουμε ε, ε, μέσα από διάφορες καταστάσεις. Δεν καθόμαστε σε φορτηγά χωρίς οδηγούς. Πρέπει να περάσουμε από αυτές τις περιοχές και τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Ε, βοηθούμε 850.000 άνθρωπους, 450.000 είναι εκτοπισθέντες, αλλά ε, μόνο τελευταίως 850 έως 950 έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του Ιντλή. Πολύ περιπλοκή κατάσταση. Τα τρόφιμα που μεταφέρουμε στο Ιντλή προέρχονται από την πλευρά τη Τουρκία. Το πώ μεταφέρουμε τα τρόφιμα και τα εμπορεύματα στη Συρία, η πρόσβασή μα είναι πολύ, είναι πολύ σφαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά αυτή την συγκεκριμένη περιοχή. Και διαπραγματευόμαστε, ενώ μιλάμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, θα πάω και εγώ τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ε, ο συντονιστής μας θέλει να κάνει μια επίγουση ε, επίσκεψη εκεί, γιατί τον ανισχύει πάρα πολύ η κατάσταση, για να μην μιλήσουμε και για το θέμα των θερμοκρασιών. Μερικοί πεθαίνουν γιατί έχουν πέσει πολλοί θερμοκρασίες, δεν υπάρχουν αρκετά αντίσκηνα, οι άνθρωποι μετακινούνται, ψάχνουν διόδους να διαφύγουν, είναι πολύ ασχήμη κατάσταση μπορούσα να μιλάω για ώρες για τη Συρία. Βοηθάμε περίπου 5-6 εκατομμύρια ανθρώπους στις γύρω περιοχές, η Ορδανία, Ιράκ, Τουρκία και Λίβανο κλπ. Κορονοϊός δεν συνειδητοποιούν πάρα πολύ ότι το επιστημικό πρόγραμμα, βέβαια το γνωρίζουν πολύ το, το παγκόσμιο επιστημικό πρόγραμμα, αλλά δεν ε, γνωρίζουν τη μεγάλη κλίμακα της ανθρωπιστικής βοήθειας παρέχεται. Αλλά όταν μιλάμε για την εμπόλα ή τον κορονοϊό, όταν φτάσει σε επίπεδα πανδημίας, ε, εμείς είμαστε ο μηχανισμός περιορισμού. Εμείς μεταφέρουμε τα υλικά, τα, τα εφόδια. Ε, ε, το λέω πολύ γενικά ομιλώντας. Αλλά είμαστε ένας μηχανισμός που ελαχιστοποιούμε τις κινήσεις των ανθρώπων της περιοχής, έτσι ώστε να βρίσκονται στις θέσεις όπου χρειάζονται στήριξη και να ελαχιστοποιούμε τις μετακινήσεις και την διάδοση των ασθενειών. Ε, υποσυτισμός, σοβαρότατο πρόβλημα. Ε, βλέπουμε με τη UNICEF σε συνεργασία. Έχουμε τεράστια συνεργασία με τη UNICEF, ε, με τον εκτελεστικό διευθυντή ή εκτελεστικός διευθύντρια έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά με εμάς και αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια ζητάμε από ευρωπαϊκές εταιρείες όπως DSM να, αντί εμείς να αγοράζουμε συγκεκριμένα προϊόντα για περιπτώσεις υποσυτισμού και να στέλνουμε στην Αφρική, ζητάμε από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να πάνε και να επενδύσουν εκεί, όπως το κάναμε και στη Ρουάντα ευρωπαϊκές εταιρείες που απασχολούν ντόπιου 600-800 ανθρώπους ε, ε, σε που εκεί δημιουργούνται και οικονομικές ευκαιρίες για τους ντόπιου ε, και δημιουργούν ειδικά προϊόντα για τα παιδιά που χρειάζονται αυτά τα ειδικά προϊόντα και ειδική βοήθεια. Και παρεμπιπτόντως αυτή τη στιγμή αγοράζουμε από την Αφρική 1,6 δις δολάρια αξίας ε, υπηρεσίες και αγαθά προσπαθώντας να τονώσουμε τις ντόπιε οικονομίες και να χρησιμοποιήσουμε τα ντόπια ε, συστήματα, ακρίδα. Έκανα ένα tweet πριν από τρεις μέρες που είπα ότι είτε πρέπει να σταλούν 76 εκατομμύρια δολάρια τώρα για να λύσετε το πρόβλημα ή 1,1 δις σε 6 μήνες για να λύσουμε το πρόβλημα σε όλη την περιοχή. Ε, εμείς δεν έχουμε 1,1 να χάσουμε. Ας προλάβουμε την κατάσταση. Η ΦΑΟ ε, ηγείται στο θέμα αυτό της καταπολέμησης ακρίδας, αλλά ε, και εμείς ε, παρέχουμε ε, εργαλεία, αεροσκάφη, προγράμματα παρακολούθησης, μετακίνηση καυσίμων, εφοδίων, ό,τι και αν χρειάζονται. Δουλεύουμε μαζί με τις αρχές στην Κένια, στην Ουγγάντα. Δεν ξέρω αν είδατε μια έκθεση, αλλά η ακρίδα τώρα έχει περάσει στο νότιο Σουδάν σε περιοχή του Ισημερινού που ε, πλήττεται και από πόλεμες καταστάσεις και από πλημμύρες. κατάσταση επιδεινώνεται με την αύξηση των ακρίδων. Ο κορονοϊός τώρα βρίσκεται στην Αφρική. Υπήρχε ένα περιστατικό στο Κάιρο. Ε, δεν μιλάω τώρα με δεικτικά στοιχεία, αλλά με πολλούς εργαζόμενους στην Αφρική. Ε, φαντάζομαι ότι η γρήπη αυτή δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει φτάσει σε μερικέ χώρε τη Αφρικής. Τώρα, αν έχει φτάσει ή όχι, δεν το ξέρουμε, αλλά αν φτάσει σε επίπεδα πανδημίας, τότε θα ενεργοποιήσουμε μια άλλη ε, επιχείρηση. Ήδη κάνουμε συναντήσεις με χώρες και έχουμε συζητήσει για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση αυτής της ενδυνάμει πανδημίας. Πολλοί έχουν ξεχάσει και τη γρήπη των πτηνών, τη γρήπη των χείρων. Ε, υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα από φωτιές, από ακρίβες, από πλημμύρες, από γρήπες που απαιτούν εξαιρετικές προσπάθειες. Ε, με τις καταστάσεις που προκαλεί ο άνθρωπος και τις κλιματικές καταστάσεις έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας το 2020. Αλλά αν είμαστε στρατηγικοί στις δαπάνες μας και στα προγράμματά μας, μπορούμε να επιφέρουμε σταθερότητα σε περιοχές όπου θα επηρεαστούν και ε, ε, όπως έλεγα, ε, μιλούσα με ηγέτες της Γερμανίας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, είπα, και τον είπα, η επιστημιστική ασφάλεια είναι κρίσιμη σημασία, έλεγα. Και όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι έχουμε λύσεις να σταματήσουμε την μετανάστευση εξ ανάγκης. Τώρα, την εξαναγκαστική μετανάστευση ε, όπου οι οικογένειες προσπαθούν να ε, εξασφαλίσουν τη διαβίωση των παιδιών τους. Τώρα έχουμε και επιπρόσθετα προβλήματα όπως η ακρίδα και οι πλημμύρες και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας και πάλι θα ήθελα να ζητήσω να μην διστάσετε να έρχεστε μαζί μας επί τόπου όταν πάτε στο, Βόρειο Σουδάν, στο Νότιο Σουδάν ε, να συναντηθείτε με τους συντονιστές μας, να δείτε τι συμβαίνει εκεί και πώς δαπανώνται επατολεσματικά τα χρήματα. Και ένα τελικό σχόλιο, και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο αίτημα που έχω από εσά. Τώρα που είμαι στο σύστημα του ΟΗΕ, ε, η μεγαλύτερη μου ανησυχία είναι ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠΑ και άλλοι δωρητές, οι διεθνείς, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι στρατηγικά. Έχω δει χώρε όπου η Γερμανία κάνει λίγο από εδώ, η ΕΠΑ λίγο κάπου αλλού, το Ενωμένο Βασίλειο παρέχει κάτι αλλού. Όχι. Αυτό δεν θα μας δώσει μακροπρόθεσμες λύσεις. Θέλουμε στρατηγικό σχεδιασμό, ολοκληρωτικό σχεδιασμό ε, ιδιαίτερα για εύθραυστες περιοχές όπως είναι η Αφρική. Αν δουλέψουμε στρατηγικά ενωμένα, είμαι ε, σίγουρος ότι θα έχουμε πιο, αποτελεσματικ... πιο, πιο μεγάλα αποτελέσματα. Ε, εγώ λέω ότι αν δεν το κάνουμε με στρατικό τρόπο θα μας κοστίσει 100-200 φορές περισσότερο εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις γεννησιουργίες αιτίε. Σας ευχαριστώ και είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε οποιασδήποτε ερωτήσεις, να εμπλακούμε και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, είναι οι σύμμαχοί μας και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες εκεί έξω στον πλανήτη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε όταν πάμε στο Σουδάν ε, και ίσως να πάμε και στο Λίβανο. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε ε, με τους συντονιστές να έχουμε και κάποια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος. Σας ευχαριστώ κύριε Μπίσλη για την παρουσία σας. Καλά περάσετε στις Βρυξέλλες.